Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Λάγκεν για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Δίνω αμέσω το λόγο στον κύριο εισηγητή, τον κύριο Λάγκεν, για τέσσερα λεπτά. Να. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, θέλω καταρχήν πρώτα να ευχαριστήσω για την συνολικά πολύ καλή συνεργασία που είχαμε σε πολλές συνεδριάσεις ε, προετοιμάσαμε τις ε, συναντήσεις ε, μας και, υπάρχουν και υπήρχαν και κάποια ανοιχτά ερωτήματα, όμως πιστεύω ότι ιδιαίτερα φιλικά για τους καταναλωτές μπορέσαμε να κατλήψουμε την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Θέλω να αναφερθώ στα πιο σημαντικά στοιχεία σε σχέση με αυτό το θέμα. Πρώτον, ότι οι καταναλωτές σε σχέση με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τα πολλά γραφεία μπορούν πραγματικά να βρουν μια πρακτική δυνατότητα ε, κάλυψης των αναγκών τους. Τα δικαιώματα των καταναλωτών και το πώς θα πρέπει να ανταμείβονται οι διαμεσολαβητές διευκολύνονται. Μια καλύτερη διαφάνεια που διασφαλίζεται ώστε τα συμφέροντα των ε, καταναλωτών να τίθενται στο επίκεντρο. Και βρήκαμε και εγκρίναμε ένα συμβιβασμό που τους ε, καλά λειτουργούντες μεσολαβητές πολίτες στην Ευρώπη πρέπει πραγματικά να δούμε ότι δεν είναι εκείνοι οι οποίοι προκαλούν κάποιες καταστάσεις που κατά τα άλλα μπορούν να αποφευθούν. Εισάγουν κάποια στοιχεία που βοηθούν τους καταναλωτές να γνωρίζουν τι γίνεται σε σχέση με τα ασφαλιστικά τους, ασφαλιστικά τους συμβόλαια, τη διάρκεια των ασφαλιστικών τους συμβολέων και το τι καλύπτουν. Και σε σχέση με τον τομέα ασφαλίσεων πανευρωπαϊκά διασφαλίζεται υπεραιτέρω ανάγκη κατάρτισης και επιμόρφωσης των ε, ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Και μέσα σε μια τακτή περίοδο, σε μια ελεύθερη επιλογή 200 ωρών, δηλαδή μια εβδομάδα ανά από ανεξάρτητους φορείς μπορεί να διασφαλίζεται αυτή η περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση των υπεύθυνων. Υπεύθυνα για αυτή την κατάρτιση επιμόρφωση θα είναι τα κράτη-μέλη. Έχουμε ένα κεφάλαιο για το οποίο συζητήσαμε διεξοδικά, που είναι τα ε, προϊόντα, τα ασφαλιστικά προϊόντα, που συμφωνήσαμε όπως και για τα MIFID μέσα στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών, ε, της χρηματοοικονομικής προσέγγισης να αντιμετωπίζονται. Παρόλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, οι, ιδιο, οι τους. Ε. Τα ίδια προϊόντα στην ασφαλιστική αγορά θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο να ρυθμίζονται. Αυτό εκάστοτε θα πρέπει να ρυθμίζεται από τα νομικά κείμενα και να μην, υπάρχουν, να μην δημιουργείται σύγχυση με κερδοσκοπικά προϊόντα τα οποία διοχετεύονται στην αγορά. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε ότι σε σχέση με την ασφαλιστική αγορά υπάρχουν διαφορετικά προϊόντα και πρέπει να διαφοροποιούμεθα στην αντιμετώπιση τους. Ε, λαμβάνουμε υπόψη αυτή τη διαφοροποίηση και προσφέρουμε στους καταναλωτές εύληπτες πληροφορίες μέσα σε ένα διαφανές πλαίσιο χωρίς να αντιμετωπίζονται αρνητικά οι μεσολαβητές. Ε, εδώ σε σχέση με την αποκάλυψη στοιχείων των συμβολέων υπάρχουν επιθυμίες να αποκαλύπτονται διάφορα ε, δεδομένα, υπάρχουν ε, και τα θέματα της ε, κάλυψης των αναγκών των καταναλωτών όσον αφορά και προϊόντα επενδυτικά. Έχουμε επίσης και την απλούστευση των συνδυασμένων δράσεων, καθώς επίσης και ξεχωριστή προσφορά που πρέπει να γίνεται σε σχέση με τους καταναλωτές για αυτά τα προϊόντα και αντιμετώπιση όπως και τα μη παρόμοιων προϊόντων. Νομίζω με όλα αυτά, αυτά τα οποία συμφωνήσαμε και τηρήσαμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ε, διαμορφώσαμε σε προτάσεις από κοινού με τους σκιώδεις εισηγητές. Και γι' αυτό θέλω ρητά να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για αυτή την ε, ε, προσπάθεια. Ακόμα και αν έχουμε κάποιες ξεχωριστές ψηφοφορίες για κάποια θέματα τροπολογιών, στο τέλος πιστεύω ότι θα υπερψηφιστεί αυτή η έκθεση από όλους. Ευχαριστώ και πάλι όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο επίτροπο κ. Μπαρνιέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα συζητάμε για αυτή την αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Ο εισηγητής κ. Λάγκεν το είπε μόλις μια ενημερωμένη επιλογή ασφάλισης μπορεί να μειώσει τον οικονομικό φόρτο για τις οικογένειες, όπως και για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι αναγκαίο να είναι κανείς βέβαιος ότι οι κίνδυνοι που μπορεί να διατρέξει καλύπτονται σωστά. με τις πρόοδους αυτής της αναθεωρημένης οδηγίας μπορεί να καλυφθούν σωστά με τη σωστή διαχείριση των κινδύνων, με την κατάργηση των συγκρούσεων συμφερόντων. Πιστεύω ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι μια αγορά που κυριαρχείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές φορές από πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρό επιχειρήσεις. Και δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς αυτής, η Κομισιόν, εγώ, επελέξαμε σε αυτή την πρόταση να διατηρήσουμε μία προσέγγιση ελάχιστης εναρμόνισης, απαντώντας έτσι στις κριτικές που ακούω για υπερβολική εναρμόνιση από την Ευρώπη. Ορίστε λοιπόν ένα παράδειγμα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά θέτει ένα πλαίσιο και αφήνει στα κράτη-μέλη την απαραίτητη ευελιξία για να προσαρμόσουν το πλαίσιο αυτό στις εθνικές ιδιαιτερότητες. Πολύ ειλικρινά θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο σας για το έργο του και για την ταχύτητα για αυτόν τον φάκελο του AMD2 και ειδικά να ευχαριστήσω τον κύριο Βέρνερ Λάγκεν για τις ικανότητές του τη σκληρή του δουλειά, και τις γνώσεις του και τους σκιώδεις ε, εισηγητές, ε, Όλοι Σμιτ, ε, Άσλε Φόξ, Γιώργιν Κρότερ και λοιπούς. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το δικό σας ρυθμό. Θα συνεχίσει τις εργασίες του τον επόμενο Απρίλιο. Εγώ επιθυμώ να επιτευχθεί συμφωνία μέσα στους επόμενους μήνες αν μη τι άλλο φέτος. Αυτή η εκθέση πραγματικά βελτιώνει τη δική μου πρόταση και οι ανησυχίες μας είναι οι ίδιες. Να υπογραμμίσω δύο σημεία. Αφενός ε, επιθυμούμε να ενισχύσουμε την προστασία των καταναλωτών. Έχετε άγει ένα ενημερωτικό έγγραφο για τα προϊόντα που δεν είναι ασφαλή ζωή, καθώς ε, και προς τις εξουσίε για, για τις ευρωπαϊκές αρχές Επίσης διασφαλίζεται ε, συνθήκες θεμητού και δίκαιο ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παρόχων ασφαλιστικών υπηρεσιών. Επιβεβαιώνεται το πεδίο εφαρμογής για τις επιχειρήσεις και τους διαμεσολαβητές έως και όσους πολλούν ασφαλιστικά προϊόντα ως βοηθητικό προϊόν και διασφαλίζεται και την ύπαρξη τόπο σύγκριση ασφαλίσεων. Τώρα για να δούμε προς το μέλλον, στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, θα χρειαστεί να μεριμνήσουμε να υπάρξει συνοχή με τα υπόλοιπα νομοθετικά ζητήματα που εξετάζονται παράλληλα αυτή τη στιγμή στη νομοθετική διαδικασία. Έχω στον... Πιστεύω ότι αυτό το θέμα σχετίζεται με το MIFID που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με το κανονισμό KIDIP που βρίσκεται σε φάση διαλόγου και με την οδηγία που σχετίζεται με τον ε, κανονισμό εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών. Υπάρχει μια συνοχή λοιπόν, μεταξύ όλων αυτών των θεμάτων και εγώ θα συνεργαστώ μαζί σας και με το Συμβούλιο μόλις αυτό ολοκληρώσει το Γενικό του Προσανατολισμό. Κύριε Ισίτα, κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, με αυτό το κείμενο επιτρέπουμε στους ασφαλιστές και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να συνεχίσουν σταθερά και με συνέχεια στις οικονομικές αγορές ε, έχοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θέτοντας την ευρωπαϊκή οικονομία σε αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη που αναμένουν οι πολίτες. Ε, αυτό το όραμα πρόδευσε πολύ καλά χάρη στις δικές σας εργασίες και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει ε, κύριο Στάιλερ, Επιτροπή Στέρχης Αγοράς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συγητές και τον κύριο Μπαρνιέ. Η έκθεση αυτή πήρε χρόνο να φτάσει μέχρι την Ολομέλεια. Ο στόχος της ε, αναδιατύπωσης αυτής ήταν η προστασία των καταναλωτών στην ασφαλιστική αγορά, η οποία είναι κατακαιρματισμένη κάτι το οποίο κοστίζει στους καταναλωτές, υπάρχουν ε, κάποιες ασυνέπειες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσει. Οπότε μπορεί να μην καταλάβουν καλά οι καταναλωτές τους κινδύνους, το κόστος και τα στοιχεία της ασφάλισης την οποία αποφασίζουν. Υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές πώληση επίσης. Όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Εγώ δεν είμαι βέβαια πεπισμένη ότι η αναδιατύπωση αυτή διορθώνει όλε αυτέ τι ανησυχίε των καταναλωτών. Εγώ θα ήθελα μια πιο φιλόδοξη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση βέβαια παρουσιάζεται από την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Επίση, είμαι πολύ απογοητευμένη που η αναδιατύπωση αυτή θέλει να αλλάξει τι εναλλακτικέ ε, μεθόδου επίλυση διαφορών, παρόλο που πολύ πρόσφατα έχει εμφασίσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πρόβλημα για χώρε οι οποίε έχουν προχωρήσει πιο πολύ, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, που υπάρχει οικονομικό όμπουτσμαν που παρεμβαίνει σε περίπτωση τέτοιων υποθέσεων. Εμείς λοιπόν θέλουμε μεγαλύτερη προστασία για τους καταναλωτές. Είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση, ιδιαίτερα όταν η υπόλοιπη Ευρώπη θέλει να προσπαθήσει να πετύχει όσο γίνεται καλύτερες προδιαγραφές και άρα χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει πιο πολύ δεν πρέπει να αναγκάζονται να πάνε πίσω τώρα. Επίσης την εναλλακτική επίλυση διαφορών θέλουμε να τη στηρίξουμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο κύριος Λένε δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Δίνω λοιπόν το λόγο στους ομιλητές των πολιτικών ομάδων για το ΕΛΚ, ο κύριος Πέλτσε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον συνάδελφο Βέρνερ Λάγκεν για αυτή την πολύ καλά ισορροπημένη έκθεση και όλοι οι εμπλεκόμενοι καλύπτονται θεωρώ με, από την πρόταση αυτή που κατατίθεται όσον αφορά την αγορά ε, ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Εγώ διαφοροποιούμε σε σχέση με τα προηγούμενα σχόλια. Πιστεύω ότι η μέγιστη προστασία παρέχεται μέσω αυτής της πρότασης για τους καταναλωτές και γίνονται σεβαστά ε, τα συμφέροντά τους ενώ ε, φυστάται η προσοχή στους κινδύνους και τον επιμερισμό τους και το γεγονός ότι οι πληροφορίες πρέπει να καταλήγουν στους ε, καταναλωτές έγκαιρα προτού υπογράψουν τέτοιου είδους συμβάσεις συμβόλαια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα αν υπάρχουν κάποια επίμαχα σημεία και συγκρούσεις ε, συμφερόντων, τα κράτη-μέλη να μπορούν να ε, δημοσιοποιήσουν, να καταλήξουν δηλαδή στην δημοσίευση, μπορούν να ε, ζητήσουν από τους ε, μεσολαβητές να δημοσιεύσουν τους όρους και τα στοιχεία με τα οποία έδρασαν. Πιστεύω ότι αν είχαμε μια παρόμοια ρύθμιση πριν από την οικονομική κρίση, θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει η οι διαμεσολαβητές να έχουν παραπλανήσει καταναλωτές όπως συνέβη στο παρελθόν προσφέροντας στους καταναλωτές προϊόντα χωρίς να έχουν ενημερωθεί όπως, πρέπει, ε, όπως έπρεπε οι καταναλωτές. Η επιμόρφωση και η κατάρτιση είναι σημαντικό στοιχείο σε αυτή την αγορά και πρέπει να έχει υποχρεωτικό, δεσμευτικό χαρακτήρα και πρέπει να επιμορφώνονται και να καταρτίζονται όπως είναι και σημαντικό να υπάρχει ένα στην, ως ιστοσελίδα προσπελάσιμο σύστημα καταχωρήσεων για να μπορούμε να εποπτεύουμε το τι συμβαίνει. Θα είναι πιο διαφανές έτσι αυτό το σύστημα, θα μειώνεται το γραφειοκρατικό βάρος ε, και η γραφειοκρατική επιβάρηση. Θεωρώ ότι είναι τόσο ισορροπημένη η έκθεση αυτή που θα έπρεπε να την υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο όσο περνά από το χέρι μας. Αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους, να υπερψηφίσουν την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα των σοσιαλιστών. Ε, Σάντσες Πρεσέντο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Επιτροπή Μπαρνιέ. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον κύριο Λάγκη και του άλλους εισηγητέ με τους οποίους συνεργάστηκα και εγώ για να πετύχουμε συμβασμού. Πρόκειται για πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ένα μεγάλο μέρος του ΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε υποστηρίξει, λοιπόν, να τηρούνται οι διεθνείς μας υποχρεώσεις και νομοθετικά και να υπάρχει ένα ισορροπημένο πεδίο εφαρμογής. Δεν συμπεριλαμβάνονται συμπληρωματικές δραστηριότητες ή περιπτώσεις κόστους κάτω από 700 ευρώ. Δεν είναι βέβαια ένα εύκολο και απλό προϊόν η ασφάλιση. Εξαρτάται κατά πολύ από προσωπικές επιλογές μεταξύ άλλων. Οπότε εδώ έχει σημασία να γνωρίζουν οι διαμεσολαβητές πολύ καλά τις περιπτώσεις και τους ασφαλισόμενους και να μπορούν να σταθούν στο ύψο τους όσον αφορά τον επαγγελματισμό τους. Πρόκειται για αποφάσεις που παίρνουν οι καταναλωτές αφού προηγουμένως έχουν σκεφτεί καλά. Γι' αυτό πρέπει να έχουν την κατάλληλη βοήθεια και να τηρούνται οι προδιαγραφές ε, ημιτ. Νομίζω ότι όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, τότε πρέπει να υπάρχουν και ποσοτικά δεδομένα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλείας και Επαγγελματικών Συντάξεων. Πρέπει να συνδυάζεται η ελευθερία της προσφοράς με την ελευθερία επιλογής από τον καταναλωτή, μέσα βέβαια σε απόλυτη διαφάνεια. Ελπίζω να εγκριθεί η πρόταση αυτή αύριο στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους φιλελευθέρους. Ο κύριος Σμιτ, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολιτικά καθόδες το ζήτημα αυτό όσον αφορά τους ε, διαμεσολαβητές στις ασφαλίσεις ε, οι ε, προμήθειες θα απαγορεύουν ή όχι. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει μια τέτοια απαγόρευση. Στη Σουηδία δεν έχουμε πρόβλεψη για τέτοια απαγόρευση. Έχουμε όμως ε, κάποια, ε, κάποια ποσοστά τα οποία εντάσσονται σε, ένα, σε μια τέτοια απαγόρευση. Πάντα θα πρέπει προς όφελος και προς το συμφέρον των καταναλωτών να δρά κανείς. Και είναι σημαντικό ότι δεν μπορεί κανείς να οδηγήσει σε μονοπωλιακού χαρακτήρα ασφαλιστικές υπηρεσίε. Τα κράτη-μέλη μπορούν να πάνε πιο πέρα από αυτή την πρόταση και μπορούν σε σχέση με τα τέλη, ε, εισφορέ εισφορές, ε, να ρυθμίζουν και να, να ε, θεσπίζουν και περιορισμού. Μπορούν δηλαδή τα κράτη-μέλη, σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι πρέπει να είναι πιο αυστηροποιημένο αυτό το πλαίσιο, να προχωρήσουν στι αναγκαίε ρυθμίσει. Και θα χρησιμοποιήσω τώρα ίσως ε, δυνατότητα χρήση γλώσσα που θα είναι πιο κατανοητή. Εδώ σε σχέση με την ευθυγράμμιση με το MIFID στην πρόταση του κ κυρίου Λάγκεν. Θα ήθελα να ζητήσω και από τον Επίτροπο και από τον κύριο Λάγκεν τι σημαίνει αυτό στην πρακτική εφαρμογή διότι από πλευρά του συναδέλφου κυρίου Γκίγκολτ που είναι και φίλος οι τροπολογίες 4 και 5 ακούω ότι δεν θα έχουν λέει καμία επιρροή στις ε, μελλοντικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά την ευθυγράμμιση, την συμμόρφωση των προτάσεων σε σχέση με τις διατάξεις MIFID. Έχω ακούσει όμως το αντίθετο επίσης. Και αν όλες αυτές τις τροπολογίες του κυρίου Γκίγκολ, την 9, 10 και την 11 της Δίκανης και τη ε, συσσωρεύσει, τότε αυτό τις νομικές διεργασίες και διαδικασίες θα τις καθιστούσε δυσχερέστερες ε, και πιο επιβαρημένες. Ε, θα ήθελα να μου πείτε, επαρκεί αυτό κύριε Επίτροπε, κύριε Λάγεν, με τις τροπολογίες 4 και 5 για να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τα προϊόντα MIFID. Είναι ουσιώδες αυτό για το πώς θα ψηφίσω αύριο σε σχέση με το άτομό μου αλλά και για την ομάδα μου πώς θα καταρτήσω τον πίνακα ψηφοφορίας για την ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους πρασίνους. Ο κύριος Γκίγκολ, ήταν λεπτό. Μάλιστα, αγαπητοί συνάδελφοι, η ασφαλιστική βιομηχανία ως επιχείρηση τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί ως ε, σκληρό καρύδι με τους λομπιίστες. Υπήρχαν προβλήματα και όσον αφορά και ε, τα κεφάλαια, τα αποθεματικά. Εδώ και χρόνια τα προϊόντα ως MIFID ε, έχουν καλύτερη αντιμετώπιση όσον αφορά τα συμφέροντα καταναλωτών από ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα. Γι' αυτό χαίρομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να ανταποκριθεί και να εξομοιώσει. Βρήκαμε μια ισορροπημένη τροπολογία, πρόταση σχέση συμβιβαστική που οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση σε σχέση με την αρχική πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα στην Ολομέλεια κατατέθηκαν κάποιες τροπολογίες, άλλες ενδυναμώνουν την προστασία των καταναλωτών, άλλες την αποδυναμώνουν, άλλες ε, αφαιρούν, άλλες προσθέτουν κάποια στοιχεία. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να λάβουν ως γνώμονα τον θεμητό ανταγωνισμό, όπως έχουμε την, ε, το αίτημα θεμητού ανταγωνισμού μεταξύ τραπεζών και τραπεζών τραπεζικών προϊόντων. Έτσι πρέπει να ισχύει ο ίδιο θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλιστικών προϊόντων. Στο τέλο, ε, οι διαπραγματεύσει στου τριμερεί διαλόγου δεν την χάνουν ε, τη σωστή ίδια αντιμετώπιση. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία για αυτή την εξομοίωση λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε αν δεν υπάρχουν αιτήματα για την διαδικασία Catch the Eye, ξαναδίνω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο διότι οι παρεμβάσει ε, παρουσίαζαν μεγάλη συνοχή, παρότι έγιναν μερικέ ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το πρότυπο προστασία των καταναλωτών, για το οποίο μίλησε η κυρία Στίνερ, είναι σημαντικό θέμα. Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό στους τριμερείς διαλόγους για να διασφαλίσουμε τη συνοχή, όπως είπα και εγώ, με τα υπόλοιπα κείμενα, χωρίς να ξεχνάμε τον πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα του τομέα των ασφαλίσεων. Συμφωνώ με την κυρία Γκαλπέλτς. Αν ε, είχαμε αυτούς τους κανόνες ε, και σε πολλούς άλλους τομείς, ε, όπως γνωρίζουν ο κ. Λάγκεν και οι λοιποί, γιατί εργαστήκαμε πολύ σε διάφορα κείμενα κανονισμών. Φυσικά αν είχαμε όλη αυτή την αρχιτεκτονική εποπτικών κειμένων ε, και κειμένων διαφάνειας, προστασίας των καταναλωτών, κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ε, πολλές κρίσεις δεν θα είχαν λάβει η χώρα. Πιστεύω και σε αυτή την περίπτωση, συμφωνώ μαζί σας, αν είχαμε αυτούς τους κανόνες πριν την κρίση, θα είχαμε αποφύγει την ασκή αμφίβολων πρακτικών που οδήγησαν ε, σε πολλά προβλήματα τους επενδυτές και τους καταναλωτές. Όπως και ο κύριος Σάντζες Πρεσέντο πιστεύω ότι όσο πιο ενημερωμένη είναι η επιλογή, αυστηρά ενημερωμένη, τόσο το καλύτερο. Και συμφωνώ μαζί του πρέπει να επιτυχούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ ελευθερίας επιλογής και προστασίας των καταναλωτών. Ο κύριος Γκίκολντ υποστήριξε το κείμενο και τον ευχαριστώ και ο κύριος Σμιτ ανέφερε ένα σημείο το οποίο παραμένει υποσυζήτηση κύριε Σμιτ η ευθυγράμμιση συνοχή με το ΜΥΦΕΔ ιδιαίτερα οι τροπολογίες 4 και 5 θα χρειαστεί να εξετάσουμε αυτές τις προτάσεις στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων Εξάλλου κατανοώ κίνητρα που οδήγησαν τον κύριο Συγητή σε αυτό το κείμενο. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Συγγνώμη που δεν μπορώ να είμαι πιο ακριβή, κύριε Σμίτη, σήμερα. Δεν μπορώ, θα χρειαστεί να εργαστώ περισσότερο με τον κύριο Συγητή στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων για να μπορώ να απαντήσω στα ερωτήματά σα με μεγαλύτερη ακρίβεια. Σα ευχαριστώ και την κατανόησή σα. Ευχαριστούμε. Ξαναδίνω το λόγο στον εισηγητή. Κύριε Λάγκεν, παρακαλώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για την αξιολόγηση του συμβιβασμού της συμβαστικής πρότασης και θέλω ρητά όλους τους κοιόδης εισηγητές να τους ευχαριστήσω. Στον συνάδελφο Σάντσες Πρεσέδο, τον συνάδελφο Όλε Σμιτ, τον Σβέν Άσλι Φόξ, Γιώργιο Κλούτερ, την κυρία Στάιλερ. Θέλω να του ευχαριστήσω όλους. Με όλη τη διαφοροποιημένη αρχική προσέγγιση είχαμε μια σωστή και δίκαια ισορροπημένη συζήτηση αναμεταξύ μας. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, κύριε Επίτροπε, δεν ήταν καθόλου γοργή η διαδικασία λήψης απόφασης. Κατά το θέρο 2012 είχε υποβληθεί η πρότασή σα πάνω από 1,5 χρόνο είχαμε που πέρασε από τότε που ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις. Δεν είναι λοιπόν ταχεία διαδικασία. Πότε θα ολοκληρώσουμε δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Δεν υπολογίζουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, ε, υπολογίζουμε στην, ε, θεωρούμε ότι θα γίνει αυτό την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Αναφέρθηκε η ε, αυστηροποίηση των, του κανόνα αποφυγής ε, συγκρούσεων. Ε, λάβαμε στην έκθεσή μας υπόψη αυτό το στοιχείο στοιχείο. Όμως, ποιες αρχές θα είναι υπεύθυνε το αφήνουμε στα χέρια των κρατών μελών να αποφασίζουν. Αυτό θεωρούμε γενικά ότι είναι η σωστότερη προσέγγιση. Εκεί όπου πάνε πιο πέρα τα κράτη-μέλη να μπορούν να το κάνουν αυτό, χωρίς να είναι αυτό γενική δέσμευση για όλους. Ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη όμως. Στον συνάδελφο κύριο Σάντσες Πεσέδο που στη διαδικασία ιδιαίτερα την, τα συνδυασμένα, την διασύνδεση των ε, ε συμβάσεων, των ε, πράξεων που συνδέουν και ο συνάδελφος Όλε Σμιτ είχε διαφορετική άποψη. Τώρα βρήκαμε ένα συμβιβασμό που πιστεύω εγώ προσωπικά ότι δίνει τη δυνατότητα συνενετικη επίλυση του προβλήματο. Ο συνάδελφος Σμιτ είπε κάτι για την απαγόρευση ε, προμηθειών. Τώρα, όπως τα έχουμε συμφωνήσει τα πράγματα είναι σωστό αυτό. Έθεσαν μια τροπολογία οι πράσινοι σε σχέση με αυτό το θέμα απαγόρευσης προμηθειών. Εδώ νομίζω ότι έχουμε μια σωστή συνετή ρύθμιση. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες 4 και 5 που αναφέρθηκαν σε σχέση με, το, με τα Μύφιλ. Αυτά που σήμερα σκεπτόμαστε να κάνουμε είναι συμπεριλαμβάνουν περαιτέρω ε, προτάσεις σε σχέση με το κείμενο. Θεωρούμε ότι αυτές είναι καλύτερες προτάσεις σε σχέση με την ε, προσωμείωση με τα MIFID. Πρέπει όμως στη διαπραγμάτευση να δούμε και τις ιδιομορφίες αυτών των προϊόντων και στις ε, διαπραγματεύσει και διαβουλεύσεις που θα είναι παρόντες και παρούσες οι σκιώδεις εισηγητές και σκιώδεις εισηγήτρες θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε <clears throat> σε σχέση με το κείμενο αυτό δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε ρυθμίσεις που δεν θα ταιριάζουν στα ασφαλιστικά προϊόντα. Και στο συνάδελφο Σβέν Γκίγκορτ που τον ευχαριστώ για το ότι στο τέλος αυτός έδωσε την έγκρισή του σε αυτό το συμβιβασμό εν τέλει Φυσικά έχει και κάποιες άλλες τροπολογίες, έχουμε και κάποιες άλλες τροπολογίες των πρασίνων ανέφερα τη μία για την απαγόρευση προμηθειών δεν μπορεί να την δεχτεί αυτή η δική μας ομάδα ομιλώ τώρα εξ ονόματος της ομάδας μου και η δεύτερη τροπολογία είναι το άρθρο 26α που εισάγεται εδώ όπου μια παρέμβαση ε, μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση συγκεκριμένων ασφαλιστικών προϊόντων. Αυτό είναι έργο των εθνικών αρχών και όχι της ΑΙΟΠΑ. Και γι' αυτό εμείς θεωρούμε ότι αυτό το τμήμα αυτής της τροπολογίας πρέπει να απορριφθεί. Εκεί που θα ήθελα όμως χρόνο να σκεφτώ και να προβληματιστώ είναι οι ρυθμίσεις για τις εξαιρέσεις. Έχουμε διαβουλεύσει στην δική μας κοινοβουλευτική ομάδα που βρίσκονται υπό εξέλιξη. Θα ήθελα να συζητήσω το θέμα και θα δούμε πως αύριο θα ψηφίσουμε ως ομάδα. Σε ε, αντιδιαστολή με τους ε, πρασίνους ε, έχουμε μια μεγάλη κοινοβουλευτική κοινοβουλευτική ομάδα που πρέπει με την ε, αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Θέλω συνολικά να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν. Ευχαριστούμε. Έχει κλείσει η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 11.30. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διατάξης έκθεση της κυρίας Γκροστέτ, τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας. Δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία εισηγήτρια.